δραστηριότητε, αντίκτυπο και προστιθέμενη αξία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση μεταξύ 2007 και 2014. Το λόγο έχει για τέσσερα λεπτά η εισηγήτρια κυρία Χάρκη. Ευχαριστώ Πρόεδρα. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους γιατί ήταν πολύ καλή συνεργασία και επικοδομητική όσον αφορά την έκθεση. Ευχαριστώ του Κιώδη και όλε τι επιτροπέ που συνέβαλαν με τι έξοχε γνωμοδοτήσει του. Θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα του συναδέλφου τη Επιτροπή Προπολογισμών, το, τον κύριο Ζων Πολντινόν. Λοιπόν, ο ρόλο μα εδώ ήταν να αξιολογήσουμε τι δραστηριότητε, τον αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία αυτού του ταμείου προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση και να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ποιε θα είναι οι προτάσει μα για αποτελεσματικότερη, αποδοτικότερη χρήση του Ταμείου και ευχαριστώ του συναδέλφου για τη συνδρομή του. Το Ταμείο αυτό είναι μικρό Ταμείο σε σχέση με το ESF ε, και είναι ένα νέο Ταμείο σε σχέση με το Κοινωνικό Ταμείο, αλλά μπορούμε τελικά να το διαμορφώσουμε και να γίνει θετικό. Σε αυτή την έκθεση προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τόσο ώστε να γίνει αποτελεσματικότερο αυτό το Ταμείο. Τι συμπράξεις μπορούν να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα για ε, τους ανθρώπους που έχασαν τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησεως. Πώς μπορούμε να διοργανώσουμε την διαδικασία τόσο ώστε να ανταποκρίνεται πιο έγκαιρα στις ανάγκες των εργαζομένων. Πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε καλύτερη αξία για τα χρήματά μας και για τους εργαζομένους και για τους φορολογόμενους Ευρωπαϊκής και μπορούμε να δαπανίσουμε αποτελεσματικότερα τα χρήματα. Πώ να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε σχετικά στοιχεία που μα επιτρέπουν να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα του Ταμείου χωρί να έχουμε υπερβολικέ απαιτήσει που επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη. Και βέβαια κάτι πιο κρίσιμο, πώ μπορούμε να βοηθήσουμε να εξασφαλίσουμε αεξατομικευμένα μέτρα, καλά, συντονισμένα, που ανταποκρίνονται στι ανάγκε του απολυμένου εργαζόμενου. Τι ούτω τρόπο πετυχάνουμε δύο πράγματα. Εκφράζουμε αλληλεγγύη προ αυτού σε δύσκολου καιρού και δεύτερον, τους βοηθούμε να κάνουν τη μετάβαση προς μια βιώσιμη απασχόληση. Ε, λοιπόν, το ταμείο αυτό, γιατί είναι διαφορετικό από το κοινωνικό ταμείο, το ταμείο αυτό λοιπόν αντιμετωπίζει κατεπίγουσες ανάγκες, βραχυπρόθεσμη προσέγγιση, ενώ το κοινωνικό ταμείο ε, είναι πιο διαθωτικής φύσεως. Έχουν και τα δύο ωφέλη. Και είναι πολύ θετικό αυτό που βλέπουμε. Είδαμε ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο σαν συμπληρωματικό εργαλείο όσον αφορά το Ταμείο Αντιμετωπίσεω των Συνεπειών τη Παγκοσμιοποίηση. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να πετύχουν συνεργασίες μεταξύ των δύο ταμείων, των διαφόρων ταμείων. Και τονίσαμε ότι οι πόροι του ESI μπορούν να είναι συμπροματικά μέτρα που ακολουθούν του τομεί υποστηριξη, προσωμιώνοντα ε, επένδυση και δημιουργία θέσεων απασχόληση. Λοιπόν, ποια είναι τα θετικά, ποια χρονοδιαγράμματα έχουν, ε, έχουν τα χρονοδιαγράμματα έχουν βελτιωθεί από προσπάθειε όλων, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Κρατών Μελών, Κοινοβουλίου κλπ. Οι αυταπασχολούμενοι συμπεριλαμβάνονται τώρα και μπορούν να υποφελούνται από την υποστήριξη ε, και είναι πολύ πιο περισσότεροι δικαιούχοι. Το ταμείο αυτό ανήκει στο σύστημα κοινή διαχείριση των ταμείων και επενώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το θέμα. Η συγχρηματοδότηση αυξηθεί στο 60%. Περισσότερα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν το EGF και η δαπάνη όσον αφορά τα εξατομικευμένα ε, ε, μέτρα έχει μειωθεί στο 35% και αυτές οι δαπάνες είναι ακόμα μικρότερες τώρα. Το ελεκτικό συνέδριο μας λέει ότι σχεδόν όλοι οι δικαιούχοι από το ταμείο αυτό μπόρεσαν να ωφεληθούν από εξατοκομικευμένα και συντονισμένα μέτρα. 50% ε, περίπου είναι το ποσοστό επανεπασχόλησης και κινούνται πιο έγκαιρα τα κράτη-μέλη. Εξακολουθώ, υπάρχουν προβλήματα. Τα κράτη-μέλη δεν χρησιμοποιούν το ταμείο αυτό πολύ συχνά και πιο κρίσιμο δεν χρησιμοποιούν πολύ συχνά την παρέκκληση. Η χρηματοδότηση έχει περικοπεί από 500 εκατομμύρια στα 150 εκατομμύρια. Η εφαρμογή και η υλοποίηση του προπολογισμού και απορρόφηση είναι 55% αλλά βελτιώνεται και υπάρχει και μια συγκέντρωση εφαρμογών όσον αφορά αυτοκινητοβιομηχανία, κατασκευαστικό τομέα και αεροναυτικό τομέα. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε διαφορετική προσέγγιση ανάλογα με τι ανάγκε και να βοηθήσουμε του απολυμμένου εργαζομένου. Άρα το Ταμείο αυτό πρέπει να σχεδιαστεί με έναν τρόπο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στι ανάγκε του. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει δημοσία να διαθέτουν όλε τι σχετικέ πληροφορίε όσον αφορά τι περιπτώσει που μπορεί να το Ταμείο και θα πρέπει να τεθούν στόχοι ποσοτική επανένταξη για να προσμετήσουμε την επιτυχία. Και τέλο, κάτι πολύ πιο σημαντικό είναι ότι το Ταμείο αυτό θα πρέπει να εγγυάται ότι δίνεται προστιθέμενη αξία για του απολυμμένου εργαζομένου και του και τότε μπορούμε να ζητήσουμε ένθερμα τη συνέχιση αυτού και την επέκταση αυτού. Κυρία το λόγο έχει Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πράγματι Η έκθεση αυτή ε, μου έδειξε ότι πολλοί ε, από τα συνδικάτα, από τους εργαζομένους, ε, από τη διοίκηση τρία πράγματα βλέπουν. Πρώτον ότι αυτό το ταμείο είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε έναν εργαζόμενο που έχει απολυθεί στη μοίρα του. Επίσης, από στεριόρια έχουμε μια άλλη λύση οι ε, επιταχυμένε διαδικασίε συνταξιοδότηση και το τρίτο, που θεωρώ ότι είναι και το πιο σημαντικό, νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να, ε, να εστιάσουμε στο προλαμβάνει και όχι στο θεραπεύει. Προτείνω λοιπόν εκ των προτέρων να, να βλέπουμε τι αποτελέσματα θα μπορούσε να έχει οι τεχνολογικές αυτές αλλαγές, ε, βιομηχανικές αλλαγές, η παγκοσμιοποίηση εν γέννη και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, λάβει υπόψη ναι, τη διάσταση αυτή. Να υποβάλει λοιπόν προτάσεις ώστε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο να μπορέσουμε να πλαισιώσουμε αυτές τις ε, επιχειρήσεις. Υπάρχουν πραγματικές προοπτικές κατά την άποψή μου, ιδίω για τις ΜΜΕ που με αυτή την πλαισίωση ε, δεν θα βρουν μπροστά τους τείχο όπως βλέπουν σήμερα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Εκ μέρους της Επιτροπής το λόγο έχει η Επίτροπος κυρία Τάισεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι συγητέ ε, και οι λοιποί ευρωβουλευτέ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους εισηγητές, ε, την κυρία Χάρκιν και τον κύριο για την προσοχή που έχουν ε, δώσει σε αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Κύριε Χάρκε, μάλιστα το 2007 ασχολείται με το θέμα. Είναι μια πολύ χρήσιμη για εμάς έκθεση, διότι παρά τις πολλές βελτιώσεις ε, του κανονισμού για την περίοδο ε, από το 2014 στο 2020, ε, που βλέπουμε και να αντανακλώνται στην καλύτερη λειτουργία του Ταμείου, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω τελειοποίηση. Το Ταμείο είναι ένα ε, μέσο που χρησιμοποιείται σε έκτακτες περιστάσει έχει ένα σημαντικό ρόλο. Και συμφωνώ ότι όπως είναι τα πράγματα με το προπολογισμό σήμερα, δεν μπορεί να είναι ένα εργαλείο παρέμβαση ε, για αντιμετώπιση προβλημάτων από τι απολύσει. Υπάρχουν διάφορα ζητήματα, επισημαίνονται και στην έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αξιολόγηση του EGF. Τα έχουμε ήδη λάβει υπόψη μας με τον τρέχοντα κανονισμό, όπως ε, για παράδειγμα για την αντιστάθμιση ε, έργων ε, που δεν έχουν προσθέμενη αξία για εργαζομένους που χάσει την εργασία τους και άλλες διαδικασίες. 41 εβδομάδες έγιναν 28 και Χαίρομαι που αναγνωρίζετε και τι προσπάθειε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναπτύξετε εποποιημένε διαδικασίε για τι αιτήσει και τη διαχείριση με βάση τι λειτουργικέ δυνατότητε ε, του ηλεκτρονικού στοιχείου ε, συστήματο ανταλλαγή δεδομένων. 3η Αυγούστου 2016 έχουμε το ε, απαραίτητο εργαλείο πλέον για την υποβολή των εκθέσεων, των αναφόρων. Το reporting λοιπόν θα βελτιωθεί όταν αυτό το σύστημα τέτοιες προφοριών θα είναι πλήρως λειτουργικό. Τα πρώτα αποτελέσματα της ενδιάμεσης αξιολόγησης ε, για την περίοδο 2014-2020 αναμένουμε λοιπόν να γίνει μέχρι τα τέλη του έτους, θα καλύπτει την τρέχουσα παρέκκληση, θα δίνει πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το Ταμείο και θα ε, βλέπουμε και τα θέματα των αιτήσεων 55 και άνω, οι δικαιούχοι 55 και άνω, ήταν τριπλάσιοι σε σχέση με αυτούς που ήταν από 15 24. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει απαραίτητη στήριξη, υπάρχουν αυτές οι παρεκκλήσεις οι οποίες επιβλέπουν, ε, επιτρέπουν να καλύψουμε τις τάσεις αυτές που βλέπουμε. Θέλουμε να βοηθήσουν περισσότερο τους νέους, ιδίω τους νέους ανέργους και από περιοχές με υψηλή ανεργία. Συμφωνούμε ότι το Ταμείο θα πρέπει να εξακολουθήσει να βοηθά αυτούς που βρίσκονται σε περιοχές πλέξιμος ε, από τη νέα πρωτοβουλία ε, μετά το Σεπτέμβριο του 2017, οπότε και λίγη η παρέκκληση. Με τα χαράς μπορώ να σας ανακοινώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χθες μόλις κατέθεσε πρόταση για παράταση της ε, παρέκκλησης αυτής στο πλαίσιο της συνδιάμεσης ε, αναθεώρησης του πολιτού συνομικού πλαισίου. Σημειώνω τις ανησυχίες σας ότι οι απολυθέντες από ΜΜΕ έχουν λιγότερες ε, πιθανότητες να στηριχθούν από το Ταμείο σε σχέση με αυτούς που απολύονται από μεγάλες επιχειρήσεις. Όμως η αίτηση συγχρηματοδότησης αυτό που έχουν απολυθεί από μεγάλε ή μικρότερε επιχειρήσει, είναι κάτι που έχει να κάνει στι εθνικέ προτιμήσει. Τα κράτη-μέλη σχεδόν κατά αποκλειστικότητα κάνουν τι αιτήσει με βάση τα κριτήρια παρέμβαση του άρθρου 4.1α. Ενώ άλλο, όπω η Ισπανία, το κριτήριο παρέμβαση του άρθρου 4.1β. 500 τουλάχιστον απολύσει από ΜΕ που ε, δραστηριοποιείται στον ίδιο κλάδο και σε κοντινές περιοχές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πρέπει να σας πω, προωθεί τις αναφορές από αματήμους, ανταλλαγές απόψεων, μεταξύ εταίρων για ανταλλαγή καλών πρακτικών και εφαρμογή των καλών πρακτικών από την έναρξη ισχύω του Ταμείου. Έχουμε και τις, ε, τους συνδέσμους, ε, contact persons που συναντώνται τουλάχιστον δύο φορέ το χρόνο, ανταλλάσσουν καλέ πρακτικέ. Θα στηρίξουμε την περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών για να μπορούμε να μάθουμε ένα από τον άλλο. Και θέλουμε να ενισχύσουμε την τάση αυτή. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε Τάισεν, για την παρέμβασή σας. Η κυρία Ιονγκέριος έχει το λόγο, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Ακριβώς σε ημέρες οικονομικής στασιμότητας και ενισχυμένης παγκοσμιοποίησης είναι απαραίτητο και σημαντικό να αναλάβουμε δράση για να στηρίξουμε εκείνους που είναι οι άτυχοι της ζωής. Εκείνοι οι οποίοι έχουν χάσει το παιχνίδι της ευημερία, που δεν μπορούν να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και την ευημερία, χρειάζονται στήριξη από το κράτος. Το Ταμείο έχει πολύ μεγάλη σημασία για να ε, απαλύνει το βάρος των κλειδονισμών. Πρέπει λοιπόν πάντοτε να παρακολουθούμε το δυναμικό ε, διατήρηση ή απώλεια θέσεων εργασίας σε διάφορες συμφωνίες που συνάπτουμε και μέτρα που λαμβάνουμε και βεβαίως να επιτρέπουμε στους ε, κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματεύονται ένα αποδεκτό κοινωνικό σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να στηριχθούν λοιπόν οι χαμένοι της ε, παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε την ε, γνώμη της Επιτροπής του Διεθνούς Διαδρίας. Ακούσουμε και την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Ο κύριος Βάλλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ stato finora uno strumento efficace. Per questo motivo è necessario che in futuro la Μας eh, κάνει να σκεφτούμε ότι πρέπει... Πρέπει να ερευνήσουμε όλα τα σχετικά έγγραφα ει βάθο και αυτό γιατί ε, θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις οικονομικές προοπτικές και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας στις ε, περιοχές που πλήττονται από τις απολύσεις και να δούμε ποια είναι τα αποτελέσματα που προβλέπονταν και αυτά που τελικά ε, υπήρξαν. Θα πρέπει να δούμε ωστόσο αν το κλείσιμο αυτών των εταιριών είναι αποτέλεσμα με την κατάσταση σε τρίτες χώρες ή σε άλλα κράτη-μέλη που ασκούν επιθετικές φορολογικές πολιτικές για να προσελκύσουν τις επενδύσεις. Είναι σημαντικό να μην γίνονται όλα μόνο και προς όφελος των εταιριών και η Κομισιόν να μπορεί να υποχρεώσει τις επιχειρήσεις που μετακινούνται εκτός Ένωσης να καταβάλουν αποζημιώσεις στους εργαζόμενους οι οποίοι απολύονται. Ευχαριστώ και τώρα εξ ονόματος Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ο κ. Ντόιτς. Κυρίες και κύριοι, ως ε, υπεύθυνος ε, για την γνωμοδότηση εξ ονόματος της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης θα ήθελα να τονίσω το γεγονός ε, ότι το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης και το το ESI έχουν, πρέπει να συντονιστούν ώστε να επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Η, πολιτική συνοχής Θα πρέπει λοιπόν να συντονιστούν ώστε να βρούμε βιώσιμες και μακροπρόθεσμες λύσεις, να επιτύχουμε συνεργασίες, ε, συνέργειες και να χρησιμοποιήσουμε τα διάφορα ταμεία. Ε, η περίοδος ε, υποβολής, μάλλον έγκρισης των Ετήσεων από το EGF, από το Ταμείο της Παγκοσμιοποίησης, ήταν 10 μήνες και αυτό είναι πάρα πολύ μακρύ διάστημα. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για την μείωση της περίοδου εξέτασης των ετήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα εξ ονόματος της Επιτροπής Δικαιωμάτων της Γυναίκας και της Ισότητας, η κυρία Μπλίνκεβιτσιούτε. Σας ευχαριστώ. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση πρέπει να δεχτούμε ότι βοήθησε πάρα πολλού ανθρώπου που έχασαν την ε, ε, δουλειά τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν πολύ σημαντική βοήθεια ε, στη μέση αυτής της οικονομικής κρίσης όπου πολλοί κόσμος απολύθηκε. Τέσσερις κλάδοι στην χώρα μου χρησιμοποίησαν την στήριξη της παγκοσμιοποίησης ο οικοδομικός κλάδος, ε, κατασκευές ε, ε, επίπλων επιπλοποιία ηλεκτρονική. Ε, επίσης, ε, να πω ότι το 1 τρίτο ε, των δικαιούχων είναι γυναίκες. γυναίκες. Βέβαια, για την ώρα το, οι τομεί οι οποίοι αποσχολούν περισσότερο άνδρες χτυπήθηκαν από την παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, θα πρέπει να επαγρυπνεί η Κομισιόν ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν παραμελούνται οι γυναίκες και ότι ε, υπάρχουν συγκεκριμένα πακέτα προσωπικών υπηρεσιών που θα ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες και καλό το κράτη-μέλη να συλλέγουν στοιχεία και επί τη βάση του φύλου ώστε να μπορούμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο οι γυναίκες εντάσσονται στην αγορά εργασίας και σε ποιους τομείς και αν βρίσκουν ποιοτικέ και ασφαλείς θέσεις απασχόλησης και αν βελτιώνονται οι ε, δεξιότητές τους. Ευχαριστώ πολύ μπορείτε να βασίζεστε νομίζω στην Επίτροπο μας. Είναι ιδιαίτερα ικανή στην υπεράσπιση των γυναικών στον χώρο εργασίας. Και περνάμε τώρα στους εισηγητές εξ ονόματος των ομάδων. Εξ ονόματος του ΕΛΚΟ, ο Σόγκορ. Ευχαριστώ. Εχθές συζητήσαμε τα θέματα των ε, πολιών θέσεων εργασία, τις υποθέσεις άλλων και άλλες. διαπιστώνουμε ότι μπορεί να υπάρχουν απρόβλεπτες αλλαγές σε αυτό το παγκοσμιοποιημένο κόσμο, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, κλεισίματα επιχειρήσεων και άλλα προβλήματα που μπορεί να πλήξουν ε, τη βιομηχανία και τους εργαζομένους μας. Γι' αυτό είναι απαραίτητο να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μαξιλάρι προστασίας για τους εργαζομένους μας. Έτσι λοιπόν το Ευρωπαϊκό Ταμείο έχει αποδείξει τη χρησιμότητά του και ιδιαίτερα έχει εξασφαλίσει τη δυνατότητα εξέλιξης εργασίας για τους λιγότερο ευνοημένους, τους πιο αδύναμους, λιγότερο καλά καταρτισμένους δηλαδή ε, εργαζομένους. Μπορούν βεβαίως να υπάρξουν πολλές βελτιώσεις για να γίνει πιο αποτελεσματικό και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε, να τη δεχθείτε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε. Ε, συμφωνώ μαζί σας. Θέλω μόνο να ρωτήσω το εξής. η διαπραγματεύσει, πολύ δύσκολες αυτές οι διαπραγματεύσεις της TTIP. Έχετε τη γνώμη ότι εξασφαλίζουν επαρκή κοινωνικά δικαιώματα ή θα καταστήσουν απαραίτητη την ανάπτυξη του δυναμικού του Ταμείου Αντιμετώπισης Παγκοσμιοποίησης. Κύριε συνάδελφε, νομίζω ότι ε, μας απασχολούν τα ίδια μελήματα στα κοινωνικά θέματα και άρα λαμβάνουμε με τον ίδιο τρόπο πρόνοια για να τα αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ εκ μέρους της ε, ομάδα των Σχεριστών και Δημοκρατών η κυρία Μαρία Ρενά. Ευχαριστώ πολύ τη Μαρία Χάρκιν για τη δουλειά της, ευχαριστώ πολύ τους συνεισηγητές, όπως και την Επίτροπο για τη χθεσινή της ανακοίνωση. Πώς θα δοθούν παρατάσεις για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Το ΦΕΜ βεβαίως το Ταμείο αυτό επιτρέπει την αντιμετώπιση των ε, προβλημάτων ε, εκείνων που έχασαν τη δουλειά τους λόγω της παγκοσμιοποίησης. Άρα σε ένα πλαίσιο παγκοσμιοποίησης όπως είναι αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε σήμερα πρέπει να ενισχύσουμε το εργαλείο αυτό, γιατί ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν και κερδισμένοι και χαμένοι της παγκοσμιοποίησης, όλο και περισσότερο χαμένοι μάλιστα. Έτσι λοιπόν ζητώ και περισσότερα κονδύλια, αλλά και ενίσχυση του επίπεδου της παρέμβασης και ενεργοποίηση της ρήτρα ε, εξαιρετικών περιστάσεων για να αντιμετωπιστούν οι ε, διάφορες ανάγκες που εμφανίζονται. Επίσης, και σε ένα βαθμό με πρόλαβε η κυρία Τάισεν σε αυτό που ήθελα να σημειώσω, γιατί είπε ότι δεν μπορεί να αντισταθμίζει εμπορικέ πολιτικέ στο Ταμείο παγκοσμιοποίηση. Ωστόσο, η πολιτική τη κυρία Μάλστρομ στη γενική πολιτική, όπω την έχει περιγράψει η κυρία Μάλστρομ, αναφέρεται ότι πρέπει να γίνεται ε, πρόσβαση, πρέπει να γίνεται ε, έκκληση στην υποστήριξη του Ταμείου για την παγκοσμιοποίηση όταν υπάρχουν προβλήματα εμπορικά. Από την άλλη, η κυρία Μάλστρο μας λέει ότι δεν προξενεί δυσμενείς ε, συνέπειες το διεθνέ εμπόριο. Είναι αντιφατικά όλα αυτά που μα λέει η κυρία Μάλστρομ. Το ίδιο είχαμε και χθε τη συζήτηση για την Αφρική ή για τη Γεωργία. Δεν υπάρχουν, λέει, δυσμενεί ε, συνέπειε για τη Γεωργία. Μα προφανώ και υπάρχουν. Εάν τι αρνούμαστε, δεν μπορούμε και να τι προλάβουμε και να τι αντιμετωπίσουμε. Εγώ λοιπόν λέω να τι αποδεχθούμε ότι υπάρχουν και να τι αντιμετωπίσουμε για να βοηθήσουμε πριν τη βιομηχανία πριν να φτάσει η ώρα να βοηθήσουμε του εργαζομένου που θα έχουν χάσει τη θέση εργασία του και πια δεν θα έχουν σωσ, σωσμό. Ευχαριστώ πολύ. Συντηρητικοί μεταρρυθμιστές, Γκέρικε. Δεν είναι εδώ. Φιλελεύθερη Δημοκρατική, Σαμπόν. Ευχαριστώ πολύ. Να σας καλημερίσω και πάλι. Τρίτη φορά βέβαια παίρνω το λόγο Φαντάζομαι ότι είναι έτσι δύσκολη αυτή η ολομέλεια. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε που είστε εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης και την κυρία Χάρκιν, την εξαιρετική εισηγήτρια. Να πω το εξή. Οποιαδήποτε συμμετρικό σοκ, οποιαδήποτε οικονομική αεξέλιξη, ε, οποιαδήποτε συγκυριακή αλλαγή, εφόσον ευεβιασμένη, δημιουργεί κάποιε μεταβατικές περιόδους. Αυτό ε, έχει μια δυναμική και θα υπάρξουν κερδισμένοι και χαμένοι. Για το TTIP που θα έχουμε πολύ σημαντικές εμπορικές αλλαγές. Ε, ε, μπορεί να υπάρξουν κάποιοι νικητές βράχη πρόθεσμα. Με το νέο κοινωνικό μοντέλο όμως τι θέλουμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε αυτούς που θα χάσουν έστω και βράχη πρόθεσμα, να τους βοηθήσουμε σε αυτή τη μεταβατική περίοδο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε λοιπόν και αυτό το ταμείο και να το ενισχύσουμε δίνοντας βάση στην ανάκτηση, στην επανένταξη, στην ανάκτηση ανάκαμψη, ιδίως για τις ε, πιο μειονεκτικές ε, περιοχές. Και βέβαια, εγώ θα έλεγα ότι Τανίνης. Να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία και οριζόντια να δούμε το πρόβλημα. Μπορεί να υπάρχει διακριτική μεταχείριση μεταξύ επιχείρησεων, μεταξύ τομέων. Πρέπει να βελτιωθεί αυτή η πτυχή. Ποτέ όμως δεν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρετηθεί της προσπάθειας ε, να βοηθήσει ε, την κοινωνική συνοχή όταν ε, η οικονομική συγκυρία σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποιοι χαμένοι. Η κυρία Μπόιλαν από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Χάρκιν ε, για την έκθεσή τη και να απεχίσω κάποια από αυτά που είπε. Είναι ένα θετικό ταμείο, το Ταμείο Μαγκοσμιοποίηση και το στηρίζει. Όμω αυτό συχνά χρησιμοποιείται για να αποζημιώσει τα το επιβαρυντικό αντίκτυπο των πολιτικών τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πολιτική αποβιομηχανοποίηση και ελεύθερου εμπορίου ε, που δημιούργησαν τι ανάγκε για την, για το Ταμείο παγκοσμιοποίηση. Αυτό έχει υποβαθμίσει τις, τα, τα, δικαιώματα, αυτό έχουν υποβαθμίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων και μέσα σε όλα αυτά συμφωνώ με την περισσότερη διαφάνεια αλλά και την αναφορά σε μια μεσοπρόθεσμη ε, ε, αναθεώρηση στα επίπεδα των κρατών μελών ώστε να εκτιμήσουν τα κρατημέλη την πρόοδο και να δουν ποια, σε ποια, πού θα πρέπει να παρέμβουν επιγόντως. Σε πολλέ χώρε όπω στην Ιρλανδία, τη χώρα μου, υπήρξε υπό απορρόφηση αυτών των χρημάτων και μάλιστα υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή των κονδυλίων. Αυτό είναι πολύ άδικο για τους εργαζόμενους που το δικαιούνται. Επίσης καλωσορίζω την αναφορά στη δημιουργία ισχυρότερων ε, σχέσεων εργασίας ε, ε, Πρόκειται για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων. Είναι καλή η έκθεση αυτή εν γέννη και ευχαριστώ και πάλι την κυρία Χάρκιν για την ε, συνένεση που διαγράφεται για την έκθεση της. Κυρία Μπόιλαν, έχετε μια μπλε κάρτα. Θέλετε να απαντήσετε. Mr. Hull, you have the floor. Thank you, uh, Έχετε το λόγο. Συμφωνώ με ο κύριο Γούλφ. Συμφωνώ με την ανάλυση σα για τα προβλήματα του EGF, αλλά δέχεστε ή όχι την αρχή ότι η ίδια η ύπαρξη του Ταμείου Παγκοσμιοποίηση επιτρέπει στο διοικητικά στελέχη των μεγάλων ομίλων να προβαίνουν σε απολύσει, γνωρίζοντα ότι μπορούν να απολύσουν ε, ελεύθερα και να ξεφύγουν με τι πολιτικέ του λόγω ακριβώ τη ύπαρξη αυτού του Ταμείου. Και αν δεν υπήρχε θα αναγκάζονταν από τα εθνικά κράτη να βάλουν τα δικά τους χρήματα και στις αποζημιώσεις των μασοναπολίων. Ναι. Συμφωνώ με τη μεγάλη πλειοψηφία των όσων είπατε. Βεβαίω, ω κάποιο που ήταν μέλο συνδικάτων για πάρα πολλά χρόνια, αυτό που με ενδιαφέρει είναι εργαζόμενοι. Και αν και πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε πολλά για να εξασφαλίσουμε σωστέ αποζημιώσει, σωστέ συλλογικέ διαπραγματεύσει για του εργαζόμενου, αλλά και να αλλάξουμε την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το εμπόριο και στις σχέσεις της με τις πολυεθνικές, ε, ε τους πολυεθνικούς ομίλους που μεταχειρίζονται τους εργαζόμενους ε, ε, κατά αυτόν τον τρόπο. Το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση είναι το μόνο που έχουμε. Το δέχομαι γιατί, είναι ότι, γιατί πρέπει, χρειαζόμαστε οτιδήποτε μπορούμε να καταφέρουμε, ειδικά στην Ιρλανδία αλλά και στα άλλα κράτη-μέλη αλλά είμαι, ε, συμφωνώ ότι πρέπει να αλλάξουμε την κατεύθυνση και τον τρόπο μεταχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, των ε, πολυεθνικών ομίλων. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας και για την απάντησή σας. Και τώρα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, η κυρία Ευχαριστώ πολύ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια κυρία Χάρκιν για την ιδιαίτερω επικοδομητική και πολύ καλά στοχευμένη και ευχαριστή συνεργασία για μας τους πράσινους. Η ευρωπαϊκή παγκοσμιοποίηση είναι ένα, το, ευρωπαϊκό μέσο για την παγκοσμιοποίηση δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο αντιμετώπισης των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης όταν κανείς χάνει τη δουλειά του ή κινδυνεύει να περιπέσει σε φτώχεια. Πρόκειται για ένα από τα λίγα εργαλεία με τα οποία μπορεί, ένα από τα λίγα εργαλεία που έχουμε για να σηκώσουμε τον ε, πολίτη, άνδρα ή γυναίκα που κινδυνεύει να πέσει στα ε, χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα. Έτσι λοιπόν θέλουμε ιδιαίτερος να επισημάνουμε πως η αξιολόγηση των συνεπειών ως προς τα ισότητα των φύλων έχει πολύ μεγάλη σημασία. Χαιρόμαστε ιδιαίτερως για το ότι έχει συμπεριληφθεί. Άρα μπορεί να αξιολογηθεί το κατά πόσον τόσο άνδρες όσο και γυναίκες αξιοποιούν αυτές ή μπορούν να υποφεληθούν από αυτά τα ε, βοηθήματα του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης. Θέλουμε πάντως το Ταμείο να μην γίνει μια έμεση πολιτική στήριξη των ομίλων ή ε, διόρθωσης λαθών της εμπορικής, διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Πρέπει να προστατεύει και να προσφέρει τη βοήθειά του σε όλους τους εργαζομένους άνδρες και γυναίκες όλων των κρατών και όχι μόνο αυτούς οι οποίοι έχουν την καλύτερη ενημέρωση πρέπει να καλύπτει και τα κενά και παραθυράκια που αναφέρθηκαν και από άλλους συναδέλφους σε ορισμένα κράτη-μέλη. Πρέπει να καλυφθούν αυτά ώστε ό,τι είναι ε, υποχρέωση του κράτους μέλους μέσα από την κοινωνική πολιτική να μην είναι δυνατόν να ε, παραμελείται για να αναλάβει δράση μόνο το Ταμείο για την Παγκοσμιοποίηση αυτά και ελπίζω ότι θα έχουμε μια καλή εξορρόπηση ανδρο, δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Ευχαριστώ πολύ Ευρώπη των Ελευθεριών και της αμείς Δημοκρατίας. Ευχαριστώ Κύριε Πρόεδρε, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση. Αυτό κι αν είναι φημισμό. Δηλαδή, η λύση σε όλα τα προβλήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιο πολλά χρήματα, πιο πολλά χρήματα, πιο πολλά χρήματα. Όχι αλλαγή πολιτική, ούτε αλλαγή ε, κυβέρνηση. Ούτε φυσικά σε καμία περίπτωση παρέτηση από το ενίο νόμισμα που τέτοια εξαθλίωση έχει προκαλέσει ε, στα κράτη του Νότου. Δεν καταλαβαίνετε όμως ότι αυτά τα χρήματα θα τα πάρετε από του φορολογούμενου που ήδη υποφέρουν. Μπορεί να αυξηθούν τα στοιχεία του ΑΕΠΑ. Στη χώρα μου όμω η παραγωγικότητα μπορεί να είναι πιο πάνω, αλλά έχουν συμπιεστεί οι μισθοί του κόσμου ε, διότι υπάρχει μια εντελώς ε, ε, άνευ ε, οποιοδήποτε ελέγχου ε, εισρωή ευθυνού εργατικού δυναμικού. Κι όμως μπορούμε να ανακτήσουμε τον έλεγχο. Υπάρχει μια δημοκρατική επανάσταση, συντελείται τώρα με τα δημοψηφίσματα, που είναι και το καθημερινό θέμα, το πιο σημαντικό σε όλα τα κράτη-μέλη. Θα γίνουν τέτοια δημοψηφίσματα. Κολουθήστε λοιπόν το ρεύμα και ορίστε εμπορικές πολιτικές που θα ε, είναι υπέρ των δικών σας ε, περιφερειών και χωρών. Γιατί εμείς εδώ ε, θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας ε, και όχι τι θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε και επίση ε, η πλειοψηφία με, δύο, με πολλά εκατομμύρια διάφορα στη Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε υπέρ της ανάκτηση του ελέγχου της εμπορικής πολιτικής. Ακολουθήστε λοιπόν το δρόμο που χαράξαμε και αφήστε να κερδίσει η δημοκρατία και οι συμπολίτε σα. La parola non εξ ονόματο τη Ευρώπη, δράση για την ελευθερία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κανονισμός είναι απόλυτα σαφές για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ε, στόχος είναι να ξαναβρούν δουλειά οι άνθρωποι αυτοί γιατί έχουν χάσει την εργασία τους λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Νομίζω όμως πως έχουμε δει το εξή. Λιγότερο από το μισό των όσων παίρνουν χρήματα από αυτό το ταμείο βρίσκουν δουλειά. Και σίγουρα αυτό δεν είναι επιτυχία. Και έπειτα υπάρχει δεν υπάρχει πλέον αυτή η κρίση παγκόσμιου τύπου. Βέβαια υπάρχει η κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της κακοδιαχείρισης της κρίσης και επειδή κάποιες χώρες επιτρέπεται ε, να περνέρθουν στην ανάπτυξη, ενώ όλες ε, όχι. Γιατί λοιπόν να ρίχνουμε και άλλα χρήματα σε αυτή την υπόθεση εφόσον δεν βοηθάει σε τίποτα. Το πρόβλημα είναι το ίδιο το Ταμείο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πάρει την εξουσία για την οικονομική, δημοσιονομική και κοινωνική πολιτική. Και αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα και πολύ κακό σημάδι βέβαια. Ευχαριστώ. Γκέρικε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χτες Ακούσαμε την ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης και είδαμε ότι η Ευρώπη δεν ασχολείται με τον άνθρωπο. Τώρα βλέπουμε ότι θα πρέπει να είναι πρότυπο για την ε, Ευρώπη το Ταμείο για την Αντιμετώπιση των Συνθεκών ε, της Παγκοσμιοποίησης. Ναι, είναι ένα μέσων το Ταμείο το οποίο υποτίθεται πως θα βοηθήσει εκείνους που έχασαν τη θέση εργασία τους λόγω της παγκοσμιοποίησης θα τους βοηθήσει να, άμεσα να μπουν ε, και πάλι στην αγορά εργασίας όταν κλείνει μια μεγάλη επιχείρηση και αντιμετωπίζονται οικονομικοί κλειδονισμοί. Ας το πούμε έτσι. Πολύ καλά. Αλλά για να σας ε, μεταφέρω από το περιοδικό Spiegel. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι που δεν τους θέλει κανένας. Και γι' αυτό εμείς πάντοτε στην ομάδα μου παρακολουθούμε με επικριτικό τρόπο τον αγώνα για αυτό το ταμείο. Πρέπει να είναι καλύτερο το ταμείο λοιπόν αυτό λέμε. Η άμεση ενίσχυση μπορεί να έχει νόημα μόνο εάν προσφέρεται κατά τρόπον άμεσο και μη γραφειοκρατικό. Αυτή είναι ακόμη η μεγάλη η μεγάλη πρόκληση για το δεύτερο ήμιση της λειτουργίας του Ταμείου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ραγανόπουλος. Η στήριξη των μαζικά απολυμμένων που θα εμπλουτιστεί από την επικείμενη απελευθέρωση των μαζικών απολύσεων από την ελληνική κυβέρνηση και το κουαρτέτο επιβεβαιώνουν διαπιστώσει τη έκθεση ότι πρώτον οι επιχειρήσεις κλείνουν είτε από ανταγωνισμό μεγαλύτερων είτε λόγω μετακίνησης σε άλλο τόπο ή κλάδο για μεγαλύτερα κέρδη με μικρότερο εργατικό κόστος αξιοποιώντας την περίφημη ελευθερία διακίνησης κεφαλαίου από το μάστριχτ δηλαδή με άλλα λόγια καπιταλισμό. δεύτερον ο φόβος των αντιδράσεων στις απολύσεις εμποδίζει τέτοιες αναδιαρθρώσεις. σαν μέρος αυτών λοιπόν το ταμείο παγκοσμιοποίησης αναλαμβάνει να τις εκτονώσει μοιράζοντας ασπιρίνες. γι' αυτό οι αιτούντες στη βοήθειά του είναι κυρίως οι εργοδότες. τα προγράμματα κατάρτισης δηλαδή επιδότηση της εργοδοσίας με το επίδομα ανεργίας των ανέργων αν καταλήγουν σε θέση εργασίας αυτή είναι πολύ χειρότερη από την προηγούμενη οι επιδοτούμενες μικροεπιχειρήσεις κλείνουν ενώ επιτίδη λιμένονται κονδύλια του ταμείου. οι ασπιρίνες δεν γιατρεύουν τον καρκίνο της ανεργίας αγώνα τώρα να μην περάσει η απελευθέρωση των απολύσεων αυξημένο επίδομα ενεργείας σε όλου για όλη τη διάρκεια τη με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγητρία κυρία Χάρκιν. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα. Μισό λεπτό κύριε Κάζα, δεν ακούμε την μετάφραση σε όλες ε, τις γλώσσες. Όχι, στα Ιταλικά δεν ακούω τίποτα. Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Εντάξει είναι τώρα, ρυθμιστεί και μπορείτε να συνεχίσετε. Έλεγα λοιπόν ε, για τη χθεσινή συζήτηση για την εταιρεία Caterpillar ε, στο Βέλγιο, που είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα για το πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Ταμείο για την Προσαρμογή. Φυσικά και πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί και αποτελεσματικότεροι και να αναλάβουμε άμεσα δράση, διότι δεν θα πρέπει να αφήσουμε ε, τους εργαζομένους ε, να μείνουν εκτός της αγοράς εργασίας ε, και να περιμένουν για πάρα πολύ καιρό. Φυσικά βέβαια υπάρχουν και επιτεύγματα, υπάρχουν θετικά από αυτό το ταμείο και τώρα αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιούν το ταμείο στο δυνατόν περισσότερο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει οπωσδήποτε, ιδίω στους δύσκολους καιρού που ζουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Ευχαριστώ. Ουλσκοκ. Το σημαντικό είναι να αξιολογήσουμε το, Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις Παγκοσμιοποίησεις για να είναι χρήσιμο για τις μικρές ε, και τις μεγάλες ε, εταιρείες. Υπάρχουν προαποτούμενα για να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτό το, ταμείο. Ωστόσο, για παράδειγμα στην Νότια Σουηδία, δεν γνωρίζουμε ακριβώς αν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το ταμείο για την εταιρεία Findus, για παράδειγμα, διότι υπάρχει μια ολόκληρη σειρά ανθρώπων που ε, απασχολούνται στον ίδιο κλάδο, θα πρέπει να δούμε αν υπάρχουν ελαφρυντικά για τις εταιρείες που εμπλέκονται σε εμπορικές ε, συγκρούσεις. Η Κομισιόν λέει πως δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, το Ταμείο σε αυτές τις περιπτώσεις. Το Κοινοβούλιο όμως λέει πως ναι. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί μια συμφωνία σε σχέση με την εφαρμογή του ε, Ταμείου. Φυσικά το συζητούμε και με την Επίτροπο για το Εμπόριο, την κυρία Μάρστρομ, η οποία εξέφρασε την ε, διαθεσιμότητά της για μια ερμηνεία τέτοιου τύπου γιατί υπάρχουν διάφορες αρνητικές επιπτώσεις μετά από ε, εμπορικές διαπραγματεύσεις και θα πρέπει να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει αυτό το ε, ταμείο και σε αυτές τις περιπτώσεις. Κυρία Γιατεμάκη, έχετε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, το Ταμείο για την παγκοσμιοποίηση έχει δώσει βοήθεια στο να ξαναγυρίσουν στο χώρο εργασίας, στο να βρουν μια διαφορετική κατάρτιση οι άνθρωποι που έχουν χάσει τη δουλειά τους. Είναι ένα καλό παράδειγμα λοιπόν και μπορούμε να διδαχτούμε από τα όσα έχει επιτύχει. Ταυτόχρονα όμως μπορούμε να είμαστε και επικριτικοί απέναντι στο Ταμείο και τη χρήση του. Γιατί πολλές φορές έχει χρησιμοποιηθεί για να αντισταθμίσει μέτρα για να αντικαταστήσει μέτρα κοινωνικής ε, ε, εξισορρόπησης που έπρεπε να είχαν λάβει τα ίδια τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, αυτή δεν είναι η δουλειά του Ταμείου για την Παγκοσμιοποίηση, είναι καθήκον των κρατών μελών να αναλάβουν τέτοιου είδου μέτρα. Και άλλα αντίστοιχα ταμεία βεβαίω ε, υπάρχουν για να βοηθούν του ανθρώπου. Εάν δείτε όμω τα ποσοστά της επανέβρεσης θέσης εργασίας που παρουσιάζονται από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης έχουμε ένα ποσοστό περί τα 40%. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια, ήταν εξαιρετική η έκθεσή της και περιγράφει με εξαιρετικό τρόπο τις δραστηριότητες του Ταμείου. Σας ευχαριστώ πολύ. Διαδικασία Catch Heckman. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Η έκθεση της ε, κυρίας Χάρκιν ε, συνοψίζει με πολύ καλό τρόπο το ότι έχει πετύχει μέχρι τώρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογή την παγκοσμιοποίηση και πράγματι είναι πολύ σημαντικό και καταδεικνύεται πόσο μεγάλη ανάγκη έχει να ε, κάνουμε τη διαφορά μεταξύ συμπληρωμα του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση, που ναι, είναι συμπληρωματικά, αλλά δεν είναι το ίδιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο πρέπει να γνωρίζουμε ότι βασίζεται σε μια μακρά περίοδο προγραμματισμού, ενώ το Ταμείο Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ad hoc, θα έλεγα, κατά περίπτωση. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε τη βέλτιστη δυνατή αποτελεσματικότητα και συνέργεια μεταξύ αυτών των δύο μέσων. Επίση, πολύ σημαντικό είναι να επενδύσουμε σε μακροχρόνιες λύσεις που θα μεταφράζονται σε πραγματική βελτίωση της αγοράς εργασίας. Δυστυχώς, εάν δούμε πόσοι άνθρωποι ε, είναι αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίε με βάση τη στήριξη από το Ταμείο, είναι πολύ λίγος ο αριθμός αυτός ακόμα. Νεκρέσκου. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να λάβω το λόγο γιατί είμαι ειδικό συζητητή των Σοσιαλιστών στην Επιτροπή των Προπολογισμών για τα κονδύλια του Ταμείου. Έχω συχνά αναλάβει ε, τις εκθέσεις και την παρακολούθηση διαφόρων διαφορών έργων και έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Πρέπει να μειωθεί το, ο αριθμός των απολυθέντων ε, για να μπορούν περισσότεροι να υποφελούνται και επίσης θα πρέπει η Επιτροπή να μεριμνήσει για μια πιο ομοιόμορφη εφαρμογή στα κράτη-μέλη γιατί κάποια κράτη-μέλη φαίνεται να χρησιμοποιούν περισσότερο από τα άλλα το Ταμείο. Χρειάζεται λοιπόν καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική από πλευρά Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα κράτη-μέλη ε, πιο αποτελεσματική επικοινωνία. Είναι ένα χρήσιμο μέσο για την καταπολέμηση της ανεργία στο Ταμείο. Πρέπει ωστόσο να βρούμε και έναν τρόπο για την κατάλληλη χρηματοδότησή του. Αποτελεί μια ταχεία ανταπόκριση στις δυσμενείς συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, ωστόσο χρειαζόμαστε και συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ κύριε Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση συστάθηκε με σκοπό την παροχή στήριξης προς τους εργαζομένους που απολύθηκαν λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών ή εξαιτίας της παγκόσμιας χρηματοοικονομικής κρίσης. Για την περίοδο 2013 ο ετήσιος προϋπολογισμός του Ταμείου ήταν 550 εκατομμύρια ευρώ. Όμως για την φετινή χρονιά το ποσό αυτό θα πέσει στα 150 εκατομμύρια ευρώ. Συγκεκριμένα το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως για τη χορήγηση βοήθειας ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ στους 557 απολυμμένους του σούπερ μάρκετ Λάρισα στην Ελλάδα, έπειτα από αίτηση που είχε υποβληθεί από τις ελληνικές αρχές στις 26 Νοεμβρίου του 2015 επομένως δεδομένου του ρόλου του ταμείου παγκοσμιοποίησης και όπως ζήτησα ήδη με γραπτή μου ερώτηση στις 26 Απριλίου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει αντίστοιχα με την αποζημίωση των απολυμμένων του σούπερ μάρκετ Λάρισα να δρομολογηθεί άμεσα και η αποζημίωση των απολυμένων από την ηλεκτρονική Αθηνών στην Ελλάδα η οποία κήρυξε πτώχευση αφήνοντας άνεργους πάνω από 500 εργαζόμενους. Ευχαριστώ. Κυρία Χάρκη, όχι, με συγχωρείτε. Πρώτα ο κύριος Τόμτ. Τόμτς. Η κυρία Τόμτς, συγγνώμη. Εγώ παρακολουθώ τι γίνεται με αυτό το ταμείο. Το παρακολουθώ, παρακολουθώ τις αλλαγές. Στις αρχές οι κανόνες ήταν εξαιρετικά άκαμπτη και το ταμείο θα ίσχυε μόνο για τις μεγάλες εταιρείες, αλλά τώρα μόνο αυτοί που αυτοποδοσολούνται μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ταμείο. Βεβαίως δεν έχουμε κάνει αρκετά σε αυτό το τομέα. Χρειάζεται να δουλέψουμε περισσότερο για την ευελιξία και την προσαρμοστικότητα. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση σε αυτό το ταμείο τουλάχιστον όχι ανοιχτή. Οι εταιρείε και τα κατημέλη χρησιμοποιούν ε, το ταμείο αυτό. Ε, με τα λύπης μου λέω ότι μόνο μία αίτηση από τη δική μου χώρα, τη Σλοβενία, ε, ε, είχε αίσια έκβαση και θα ήθελα να δοθεί περισσότερη δημοσιότητα στο τι γίνεται στο ταμείο αυτό, ώστε να μπορεί ο κόσμο να έχει πιο εύκολα πρόσβαση. Μάλιστα, φτάνουμε στο τέλος της συζήτηση. Πρώτα η Επιτροπός Τάισεν και μετά η εισηγήτρια Χάρκιν. Κυρία Τάισεν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί ε, κύριοι βουλευτές, να εκφράσω ακόμη μια φορά την εκτίμησή μου για την εργασία της εισηγήτριας και επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο εξ ονόματος της Επιτροπής για τις πολύτιμες προτάσεις του για περαιτέρω βελτίωση της ε, λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και της προσπάθειας να προσαρμογήσει στην ε, προσαρμογή στις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας ε, όσο το επιτρέπουν οι κανόνες και η νομική βάση. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, αλλά έχει σχεδιαστεί το Ταμείο αυτό, ώστε να αντιδράσει σε συγκεκριμένες ε, περιστάσεις όπως ε, το κλείσιμο κάποιων κλάδων. Προσωπική μου άποψη είναι ότι η πρόληψη είναι πάντοτε καλύτερη από την διόρθωση των ζημιών. Γι' αυτό και η εμπορική πολιτική θα πρέπει να συνοδεύεται από την κοινωνική και τη βιομηχανική ώστε να προετοιμάσει τις οικονομίες μας για τις αλλαγές που ε, πυροδοτούνται και από άλλους εμπορικούς εταίρους. Σύμφωνα με τις ε, εμπορικέ μας συμφωνίες ε, έχουμε και αξιολόγηση επιπτώσεων ως ρήτρα. Θα πρέπει μια εμπορική συμφωνία να ωφελεί και, τους δύο, τα δύο μέρη. Ωστόσο δεν μπορούμε να αποφύγουμε ε, ότι κάποιοι τομείς της οικονομίας μα θα υποφέρουν. Συμμερίζομαι τις απόψει τη Εσυλία Μάλστρομ ότι κάτι πρέπει να γίνει ώστε να αντιμετωπίσουμε πιθανά ε, σε αρνητικές επιπτώσεις ε, σε ορισμένου τομείς και το ταμείο σε αυτό το σχεδιασμό, το σημερινό σχεδιασμό δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Αξιότιμοι κύριοι Ευρωβουλευτέ, θέλω να σας διαβεβαιώσω, να σα καθησυχάσω ότι όπως είπε και ο Πρόεδρός σα, θα εξασφαλίσω, θα μεριμνήσω ότι όλες οι πολιτικές, για όλες τις πολιτικές θα ε, υπάρχουν και θα χρησιμοποιούνται οι δείκτε περί φύλου και περί ισότητα. Και επίσης Βεβαίως θα πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο τις ιδέες της έκθεσης και να προετοιμάσουμε τη νομική βάση για τη λειτουργία του EGF πέρα από το 2020. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Ευρωβουλευτές. Και εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα η συγγήτρια, η κυρία Χάρκιν. Πρόεδρε, ευχαριστώ, ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση δεν θα καταστεί δυνατόν να απαντήσω σε όλες τις παρατηρήσεις θα ε, αναφερθώ όμως ως δυνατόν περισσότερες είπατε εσείς ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το Ταμείο ε, Απόλυης Θέσεων που προκύπτουν κατόπιν εμπορικών συμφωνιών το, ε, απαντήσαν όμως ορισμένοι συνάλφοι κυρίως η κυρία Ρενά η οποία είπε ότι η Επίτροπος Μάλστρομ είχε αναφέρει νωρίτερα ότι θα μπορούσαν μέχρι και 150 εκατομμύρια να ε, στηρίξουν τις θέσεων εργασίας που προκύπτουν κατόπιν εμπορικών συμφωνιών. Πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε ανοίγοντα το βλέμμα και τον ορίζοντα εάν υπάρχει δυνατότητα με προληπτική δράση να προλάβουμε το κακό. Κάποιοι λένε ότι το Ταμείο ε, μπορεί να αξιοποιείται από κάποια κράτη για να ε, απαλλαγούν από τις δικές τους εθνικές και κοινωνικές υποχρεώσεις. Όχι, πρέπει πάντοτε να γίνεται η, βεβαίωση, πρέπει πάντοτε να δίνεται η βεβαίωση ότι τα κράτη έχουν τηρήσει τις διατάξεις εσωτερικές και αναλάβει τα δέοντα ε, μέτρα. Πάντως δεν απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στα κράτη το Ταμείο, απλώς αποτελεί ένα μηχανισμό αλληλεγγύης για τον εργαζόμενο και όχι για τον εργοδότη. Επίσης περιμέναμε ότι θα καταθέτατε πρόταση για την επέκταση της εξαίρεσης για τον ΝΙΤΣ. Δεν έχουμε μπορέσει ακόμα να αξιολογήσουμε βέβαια τις συνέπειες αυτού γιατί είναι σχετικά πρόσφατο μέτρο, μέτρο αλλά θα θέλαμε να βεβαιωθούμε ότι το ΝΙΤΣ ε, έχει μέτρα τα οποία ε, επιτελούν το σκοπό για το οποίο έχει σχεδιαστεί και όσο δυνατόν ε, πρέπει να βελτιώσουμε τη συμμετοχή σε αυτό. Επίσης αναφερθήκατε στο 1α και β, αλλά και το 2 επίσης, ε, όπου έχουμε από μικρές αγορές εργασίας αιτήσει. Ε, θέλω να ρωτήσω μήπως υπάρχει κάποια μεροληπτική στάση εις βάρος αυτών των μικρότερων περιπτώσεων, των μικρότερων επιχειρήσεων που κλείνουν κτλ. Γιατί δεν έχουμε αρκετές αιτήσει μήπως υπάρχει κάποιο ένα κενό το οποίο πρέπει να καλύψουμε. Πρέπει πιστεύω να βελτιωθεί το Ταμείο ε, και να, ε, να στοχεύσει καλύτερα τους στόχους του. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Χάρκιν για τη δουλειά.